Um, Καλή σας μέρα. Ας αρχίσουμε. Πιέζει ο χρόνος. Έτσι κι αλλιώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τη διάσκεψή της για την οικονομική σταθερότητα. Έχουμε και εμείς τη συνεδρίασή μας Και μετά από αυτήν υπάρχει άλλη. Οπότε το Κοινοβούλιο δεν θα εκπροσωπηθεί στην διάσκεψη αυτή γιατί πρέπει να είμαι και εδώ στην ε, Προεδρία. Για να μην καθυστερήσουμε άλλο, θα ζητήσω από τον Επίτροπο να επικεντρωθεί στο δεύτερο τμήμα της ομιλίας του. Θα κυκλοφορήσουμε ολόκληρη την ομιλία, αλλά δεν χρειάζεται το πρώτο τμήμα που είναι το πλαίσιο. Ας μπούμε κατευθείαν στο θέμα που μας απασχολεί σήμερα, τα μακροοικονομικά ζητήματα. Και όταν φτάσουμε στις ερωτήσεις, παρακαλώ μην ρωτήσετε για την Κύπρο. Αν ρωτήσετε για την Κύπρο, εγώ θα επιτρέψω στον Επίτροπο να πει μόνο εφόσον επιθυμεί, ότι έχει να κάνει με τα μακροοικονομικά. Τα υπόλοιπα μπορεί να τα σημειώσει και να συζητηθούν στην ακρόαση που θα έχουμε 8 Μαΐου. Οπότε οι απαντήσεις που θα πάρετε ίσως είναι μερικές. Ε, σας το λέω για να ξέρετε ότι αν ε, ρωτήσετε για την Κύπρο, αυτό θα γίνει. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Σάρων κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Καταρχάς, ε, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι και σήμερα ενώπιόν σας για τον οικονομικό διάλογό μας, για να συζητήσουμε τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και θα ακολουθήσω το αίτημα ή τις οδηγίες της και θα ασχοληθώ με το θέμα των μακροοικονομικών ανισορροπιών. θα ασχοληθώ με τα πορίσματα των σε βάθος επισκοπήσεων ή εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων που η Επιτροπή παρουσίασε πριν από δύο εβδομάδες που είναι ουσιώδες στοιχείο της ενισχυμένης οικονομικής μας διακυβέρνησης. Δεν θα ασχοληθώ τόσο πολύ με τις διαδικασίες, αλλά περισσότερο με θέματα πολιτικής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ιδιαίτερα πολιτικό θεσμικό όργανο και οι μακροοικονομικές ανισορροπίες ε, καλούν για να υπάρξει μια πολιτική συζήτηση για τις κατευθύνσεις των πολιτικών μας. Νωρίτερα, ε, τον Απρίλιο, παρουσιάσαμε τις ε, βάθος επισκοπής για 13 χώρες μέλη. Οι προκλήσεις που αναλύσαμε και συζητήσαμε σε αυτές τις βάθος επισκοπήσεις τείνουν να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Μερικά θέματα πολιτικής είναι κοινά για διάφορες χώρες τα εξή. Πρώτον, η εξωτερική προσαρμογή και των τρεχουσών συναλλαγών και του εμπορικού ισοζυγίου προχωράει, αλλά οι εξωτερικές χρηματοοικονομικές ε, υποχρεώσεις παραμένουν κίνδυνος για διάφορες χώρες. Δεύτερον, η ανταγωνιστικότητα και διαρθρωτική και κόστους παραμένει μια ζωτική ανησυχία για μια σειρά η οικονομίες της Ένωσης. Τρίτον, η απομόχλευση προχωράει στον ιδιωτικό τομέα, αλλά τα επίπεδα χρέους παραμένουν υψηλά. Αυτό σημαίνει χαμηλή κατανάλωση και επενδύσεις, οπότε παίζει αρνητικό ρόλο για την οικονομική ανάπτυξη. Και τέταρτον, οι αγορές κατοικιών προσαρμόζονται αλλά έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο να διανύσουμε σε διάφορες χώρες. Συμπέρασμα. Υπάρχουν μακροοικονομικές ανισορροπίες σε όλα τα κράτη-μέλη για τις οποίες ε, εκπονήσαμε αυτές τις βάθος επισκοπήσεις, αλλά η φύση και η σοβαρότητά τους διαφέρουν. Για την ε, Σλοβενία και την Ισπανία θεωρούμε ότι αυτές οι ανισορροπίες είναι υπερβολικές. Στη Σλοβενία όπου η οικονομική κατάσταση είναι ακόμη διαχειρίσιμη, υπάρχουν υπερβολικές μακρονομικές ανισορροπίες, οι οποίες ε, ε, πρόσφατα αυξάνονται. Σε ένα πλαίσιο αρνητικών οικονομικών τάσεων, οι κίνδυνοι για την οικονομική σταθερότητα που προκύπτουν από την υπερχρέωση των επιχειρήσεων και την απομόχλευση είναι ουσιώδης. Αυτοί οι κίνδυνοι ε, επιδεινώνονται από περιορισμένη δυνατότητα προσαρμογών στην αγορά εργασίας και τις κέφαλοι αγορές και λόγω μιας οικονομικής δομής όπου κυριαρχεί η κρατική ιδιοκτησία. Στη Σλοβενία πάντα. Για την Ισπανία. Παρά την σημαντική πρόοδο πέρυσι, το 2012, υπάρχουν ακόμη υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες πολύ υψηλό ε, χρέος των οικοκυριών, αλλά και εξωτερικό που εξακολουθεί να θέτει κινδύνους για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την οικονομική σταθερότητα. Υπήρξαν βελτιώσεις στην ανταγωνιστικότητα και σαφείς προσαρμογές των ροών, ιδιαίτερα όσον αφορά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, παραμένουν προκλήσεις τρομερές. Πολύ ψηλή ανεργία, και ιδιαίτερα ε, σφιχτές ε, συνθήκες χρηματοδότησης καταδεικνύουν ε, το πόσο ευάλωτη καθιστά την οικονομία η κατάσταση αυτή ανισορροπιών. Η Επιτροπή από κοινού με τις κυβερνήσεις της Σλοβενίας και της Ισπανίας καθώς και με άλλες κυβερνήσεις των κρατών μελών προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Θέλουμε να στηρίξουμε αυτές τις χώρες στις προσπάθειες μεταρρυθμίσεων που κάνουν και στην αντιμετώπιση των ανισορροπιών. Στην περίπτωση της Σλοβενίας, για να στραφεί αυτή η αρνητική τάση, η χώρα θα πρέπει να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησε και να συμπεριλάβει συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής στο ε, επερχόμενο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και σταθερότητας. Με τον ίδιο τρόπο η Ισπανία πρέπει να διατηρήσει το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων συμπεριλαμβάνοντας συνολικές και συγκεκριμένες πολιτικές στο πρόγραμμά της ε, μεταρρυθμίσεων και σταθερότητα. ε, συγγνώμη, προσεχώς, συγκεκριμένα αύριο, ο Πρωθυπουργό Ραχόη, μετά το Συμβούλιο Υπουργών, ελπίζουμε, περιμένουμε να υποβάλει αυτά τα, τα προγράμματα και να τα δημοσιοποιήσει. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή θα εξετάσει από κοντά τα επερχόμενα προγράμματα σταθερότητας και μεταρρυθμίσεων όλων των κρατών μελών της Ένωσης. Και μετά από αυτό οι συστάσεις πολιτικής μας θα δοθούν που θα συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο των ε, ειδικών για κάθε χώρα συστάσεων που θα υποβάλουμε τέλη Μαΐου. Συγκεκριμένα 29 Μαΐου. Το πακέτο αυτό θα καλύπτει και τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, αυτή η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και η δημοσιονομική πολιτική έχει συζητηθεί ιδιαίτερα και έντονα το τελευταίο δεκαπενθήμερο και θέλω να τονίσω την κοινή οικονομική στρατηγική της Ένωσης για να προωθήσει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να περιορίσει την αύξηση του χρέους. Για να επιτύχουμε αυτούς τους ε, διτούς στόχους ενθαρρύναμε την εξορρόπηση των δημοσιονομικών με μια συνεπή δημοσιονομική πολιτική ε, μέσο πρόθεσμα. Γι' αυτό το λόγο επεκτείναμε τις προθεσμίες για την προθεσία ε, υπερβολικού ελλείμματος για την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα πέρυσι. Με βάση λοιπόν αυτή την πολιτική μας για τα δημοσιονομικά, ο ρυθμός, ε, η ταχύτητα της δημοσιονομικής εξυγίανσης επιβραδύνεται στην Ευρώπη. Φέτος η διαρθρωτική δημοσιονομική προσπάθεια θα είναι 0,75 του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Αυτό είναι το μισό του περσινού που ήταν 1,5%. Η διαρθρωτική προσπάθεια πέφτει από το 1,5 στο 0,75 του ΑΕΠ. Που ήταν πέρυσι 1,5 λοιπόν. Οι αποφάσεις που οδήγησαν σε αυτή τη μείωση έγιναν πέρυσι με βάση, με τις, με βάση τις συστάσεις της Επιτροπής ε, το περασμένο, την περασμένη άνοιξη. Αν συγκρίνουμε με τις ΗΠΑ βλέπουμε ότι μειώνουν το έλλειμμά τους ε, κατά 1,75% φέτος. Χωρίς όμως μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική. Αυτό σημαίνει ότι σε σχέση με την ΕΠΑ φέτος εμείς κάνουμε το μισό. θα αναρωτηθείτε τι μας επέτρεψε αυτήν ε, την ε, επιβράδυνση της πορείας της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Τρεις παράγοντες το καθιστούν δυνατό. Πρώτον, η αυξανόμενη αξιοπιστία της δημοσιονομικής πολιτικής ε, της Ευρωζώνης και των κρατών που επετεύχθη από το 2011. Δεύτερον, η αποφασιστική δράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να σταθεροποιήσει τις αγορές. Και τρίτον, οι μεταρρυθμίσεις της ε, οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης που μας δίνουν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για να διαφοροποιήσουμε την ε, δημοσιονομική προσαρμογή και να προωθήσουμε τις διαθροτικές μεταρρυθμίσεις. Οι παράγοντες αυτοί μας έδωσαν ε, την δυνατότητα η δημοσιονομική μας πολιτική να έχει πιο μέσοπρόθεσμη εστίαση. Αυτό δεν ήταν δυνατόν το 2010-2011 διότι τότε ε, διάφορες ε, ε, χώρες της Ευρωζώνης κινδύνευαν είτε να καταστούν αφαιρέγγιες είτε να πέσουν στη δίνη απαγορευτικών επιτοκίων. Εκείνη τη στιγμή πολλά κράτη-μέλη έπρεπε να ξανακερδίσουν την αξιοπιστία της πολιτικής τους με πολύ δύσκολες αποφάσεις για να επανέλθει η δημοσιονομική τους πολιτική σε βιώσιμη κατάσταση. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, ε, καταλαβαίνω ότι έχει λήξει ο χρόνος μου. Να πω λοιπόν ότι είμαι διατεθειμένος να συζητήσω και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη, όπως, για παράδειγμα, ιδιαίτερα σκληρές, ε, σφιχτές συνθήκες ε, δανειοδότησης. Αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο αυτή τη στιγμή για να επιτευχθεί ανάπτυξη ιδίω στη Νότια Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν αυτή η παγίδα ρευστότητα, που είναι παγίδα χρηματοδότηση. Είναι ουσιώδε λοιπόν όλες οι προσπάθειες όλων των θεσμικών οργάνων τη Ένωση, όλων των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν αυτή, αυτό το πρόβλημα ω επίγουσα προτεραιότητα ούτω ώστε οι επιχειρήσει που μπορούν να εξάγουν και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόληση, να έχουν την αναγκαία χρηματοδότηση για να στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και προσβλέπω στις ε, παρατηρήσεις και συστάσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ερωτήσεις. Πέντε λεπτά. Ξέρουμε από πριν ποιοι θα είναι, δεν χρειάζεται να μου κάνετε νόηματα. Αλλά προσπαθήστε να τηρήσετε το χρόνο σας, γιατί αν το ξεπεράσετε τότε οι συναδελφοί σας δεν θα μπορέσουν να έχουν το χρόνο που δικαιούνται και δεν θα μπορέσουμε να συζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Διοργανική Συμφωνία. Οπότε να μην ξεπεράσουμε το χρόνο μας παρακαλώ. Ζαν Πολ, είσαι ο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ίσως από τα λατινικά να μην ε, μεταφράζεται, αλλά πάντως καταλαβαίνετε λίγο πολύ. Θέλω να σας πω κάποια σκληρά πράγματα. Τι σκέφτονται οι συμπολίτε μας σε δύσκολες περιόδους, καταλαβαίνετε γαλλικά, δεν φοράτε ακουστικά, αλλά καταλαβαίνετε. Λοιπόν, σε δύσκολες περιόδους στην πολιτική χρειάζεται θάρρος και πεποίθηση. Και έχω την αίσθηση ότι τους τελευταίους μήνες λείπουν αυτά τα δύο στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θάρρος θα ήταν να λάβουμε υπόψη μας τους καιρούς που ζούμε. Δηλαδή, η πολιτική που προτείνει η Επιτροπή είναι σωστή και να τη συνεχίσουμε ή τελικά ήταν εσφαλμένη και πρέπει να την αλλάξουμε. Αλλά το να προσπαθούμε να κάνουμε ποιότερα τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη ληφθεί είναι ένα κακό σήμα που δίνουμε. Βέβαια, βρίσκεται όλες τις εξηγήσει ότι δεν πάμε τόσο γρήγορα ως οι Ηνωμένε αλλά είμαστε καλύτεροι, έχουμε μεγαλύτερη εξοπιστή κτλ. κτλ. όλα αυτά είναι λόγια, κύριε Επίτροπε η πραγματικότητα είναι άλλη. Και αν υπάρχει μια χώρα που πρέπει να προσέξουμε όλος ιδιαίτερος, δεν είναι η Σλοβενία. Είναι μια άλλη χώρα που εγώ γνωρίζω πολύ καλά. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ξέρω αν ο κύριος Μπαρόσο έχει όντως πάρει επιστολή από τον Υπουργό των Γερμανό Οικονομικών που του παρουσιάζει τα στοιχεία τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη ιδιαίτερα στις συστάσεις όσον αφορά τη Γαλλία. Η επιστολή αυτή δεν είναι ε, μυστική, εφόσον ο κύριος Μοσκοβιτσί έχει αντίγραφο. Οι Γερμανοί συνάδελφοί μας είναι πολύ ευθύς, δεν κρύβουν τίποτα. Λοιπόν, είναι ανησυχητική αυτή η κατάσταση. Αυτά που είπε ο κύριος Μπαρόζο, που προσπάθησε έτσι να ησυχάσει τα πράγματα, τα οποία ερμηνεύτηκαν ίσως κάπως άσχημα, σχετικά με την πολιτική λιτότητα, με κάνουν πάντως να πιστεύω ότι και πάλι προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο. Την πολιτική λιτότητα τη γνωρίζουμε, πάρα πολλέ χώρε τη γνωρίζουν, υπάρχει και μια χώρα η οποία δεν τη γνωρίζει, γνωρίζει μόνο το φορολογικό περιορισμό. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να δράσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν συζητήσαμε το πακέτο των 6, των 2 κτλ, θελήσαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει στα χέρια τη τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορέσει να δράση, τουλάχιστον η πλειοψηφία. Αλλά αυτή η εργαλειοθήκη, κατά κάποιο τρόπο, που δώσαμε, τελικά παραμένει κλειστή. Και προσπαθούμε να διευθετήσουμε τα πράγματα αλλιώ. Και όχι με αυτή την εργαλειοθήκη που εμεί φτιάξαμε και περάσαμε εδώ. Γιατί δεν υπάρχει το θάρρο. Μπορεί να σα φαίνονται σκληρά τα λόγια μου, αλλά βλέπετε δεν θα ήθελα, όπω είπα και στην Ολομέλεια για την Κύπρο, σε λίγο καιρό να λέω ότι ο λόγος που οδηγηθήκαμε εκεί που οδηγηθήκαμε ήταν ότι έλειπε το θάρρος από την Επιτροπή, και εδώ δεν μιλάω για την Κύπρο, επειδή άφησε η Επιτροπή να συνεχιστούν κάποιες αρνητικές τάσεις. Θα μπορούσατε λοιπόν να με καθυσχάσετε, να μου πείτε ότι έχω άδικο. Μακάρι, αυτό περιμένω, αυτό θα ήθελα. Να μου πείτε ότι υπάρχει το θάρρος και υπάρχει και η πεποίθηση. Αυτό περιμένω να μου πείτε. Ο κύριος Ρεν. Ευχαριστώ πολύ για τις σκέψεις και τα σχόλιά σας. Για τη δημοσιονομική πολιτική είπα ότι συνεχίζουμε με συνοχή την ε, πολιτική μας της δημοσιονομικής εξυγένσης. Με συνοχή, με συνέπεια. Και για την ε, ανάπτυξη και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Συγχρόνως διασφαλίζουμε υψηλό ε, δράσεις για το υψηλό έλλειμμα που έχουμε στην Ευρώπη. Αναφερθήκατε εσείς σε κάποιες χώρες. Θα διαφωνήσω με κάτι που είπατε. Πιστεύω ότι η Σλοβενία είναι σημαντική χώρα. Όλες οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικές. Και το συμπληρώνω αυτό αναφερόμενος και σε μια άλλη χώρα που είπατε ότι γνωρίζετε καλά, τη Γαλλία. Είναι ορθό ότι η Γαλλία αντιμετωπίζει μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι το οποίο απαιτεί πολιτικές δράσεις. Ιδιαίτερα επειδή το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών επιδεινώνεται. Μετίες είναι και λογικός τους αλλά και άλλοι. Επιδεινώνεται λοιπόν αυτή η κατάσταση και άρα πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα του εξωτερικού χρέους. Γιατί μπορεί να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες όσον αφορά τη λειτουργία της γαλλικής οικονομίας και βέβαια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, μια που η Γαλλία είναι μια σημαντική χώρα ε, οικονομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σταματήσετε εδώ. Η Ελίζα Φερέρα έχει τώρα το λόγο. Κύριε Επίτροπε, Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που εφάρμοσε κατά γράμμα τις προσταγές της Τρόικας. Μας είπαν στην Πορτογαλία ότι αν ακολουθήσουμε όλες τις συστάσεις, τότε θα ξεφύγουμε από την κατάσταση του 10 το 10 είχαμε ένα χρέος του 93% του ΑΕΠ. Μετά τις συστάσεις σήμερα βρισκόμαστε σε 124% χρέος έναντι του ΑΕΠ. Είχαμε ανεργία 13%, σήμερα έχουμε 19%. Έχουμε 18,8% που τίνει προς το 19%. Σύμφωνα με αυτά που μας λέει η Τρόικα θεωρήσαμε ότι το 2013 θα είχαμε ένα ρυθμό ανάπτυξης. Όμως υπάρχει φθήνουσα πορεία κατά 3,2 πέρσι και 2,3 φέτος. Φτάνει, φτάνει κύριε Επίτροπε, φτάνει αυτή η συνταγή. Εγώ σήμερα είμαι πολύ απογοητευμένη διότι περίμενα ότι μετά τις δηλώσεις της Επιτροπής η οποία ανέφερε ότι η λιτότητα έφτασε στα όρια της υπό πολλές πτυχές και για να είναι μια πολιτική επιτυχής πρέπει και να συνταχθεί σωστά αλλά και να τύχει οικονομικής και κοινωνικής υποστήριξης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξετε άρδιν τις πολιτικές σας. Εσείς επιμένετε, αλλά όταν μια πολιτική δεν είναι λειτουργική, τότε θα πρέπει να πω ότι μόνο οι μοροί δεν αλλάζουν στάση, όπως λέμε εμείς τα πορτογαλικά, για να μην το πω και πιο βαριά. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να μας οδηγήσετε στον όλεθρο. Και αυτό αφορά και τον πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος είναι υπόλογος. Αλλά αυτό το βάρος θα επιβαρύνει τους πολίτες που δεν φέρουν και καμία ευθύνη. Σας ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Φερέιρα. Σε σχέση με την Πορτογαλία θα θυμόσαστε πολύ καλά ότι η Πορτογαλία είχε να κάνει με άτακτη χρεοκοπία. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποφάσισαν να βοηθήσουν την Πορτογαλία για να αποφευχθεί αυτή η άτακτη χρεοκοπία και να φτάσει σε μια οικονομική αποκατάσταση και σταθερότητα, ιδιαίτερα ως προς τα δημοσιονομικά της. Γνωρίζω πλήρως ότι αυτή η προσαρμογή ήταν επώδυνη για τους πολίτες πολλών χωρών που αντιμετωπίζουν μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Αυτό τονίζει και τη σημασία ανάσχεσης αυτής της κρίσης με συνεκτικές πολιτικές και συνεπείς πολιτικές, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να αποκαταστήσουμε τα θεμέλια της οικονομικής ανάπτυξης και να βελτιώσουμε την απασχόληση. Γι' αυτό η δημοσιονομική εξυγείωση θα πρέπει να είναι φιλική προς την ανάπτυξη και κοινωνικά δίκαιη για να είναι αποδεκτή από τους συμπολίτες μας. Αυτό είναι ύψης της σημασίας και καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλη πρόκληση για όλες τις χώρες οι οποίες βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία της δημοσιονομικής επανισορρόπησης και την χάνουν υποστήριξη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την ε, Επιτροπή και την ε, Τρόικα. Και εδώ μιλάω για την Ιρλανδία, την Κύπρο και την Πορτογαλία που βρίσκονται σε αυτή την πολιτική. Η κυρία Φερέιρα χωρίς... Ε, δεν έχει ε, μικρόφωνο. Σας λέμε μόνο μπάστα, αρκεί. Δεν χρειάζεται καν να βάλετε τα ακουστικά σας κύριε Επίτροπε. Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι σχόλιο, λέει η Πρόεδρος. Επόμενη ερώτηση από τον κύριο Κλίντς, από τους φιλελεύθερους. Κύριε Επίτροπε, είπαμε ότι είναι ανάγκη να υπάρξει ανάπτυξη. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ανάπτυξη. Με εκπλήση. ότι η Κομισιόν δεν λαμβάνει υπόψη κάτι που θα μπορούσε εν μέρη να οδηγήσει σε ανάπτυξη. Δηλαδή να ολοκληρώσει την εσωτερική αγορά στον τομέα των υπηρεσιών και να μειώσει ριζικά τη γραφειοκρατία. Η Κομισιόν για χρόνια τώρα λέει ότι πρέπει να καταργηθεί η γραφειοκρατία, αλλά όπου και να κοιτάξουμε αυτό το τέρας αυξάνεται στην, στις Βρυξέλλες. Δεύτερον, η πολιτική σας, όπως το είπε και η Ελίζα, η πολιτική σας λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν πια καμία ευθύνη. Γίνονται σαν ανήλικες. Εμείς πρέπει να δώσουμε ευθύνες στις ε, χώρες. Οι χώρες που, οι οποίες αναλαμβάνουν την τύχη τους, σκεφτείτε τι έγινε με τη Λετωνία. Το 1999 έλαβε μέτρα, ενώ ήταν σε μια τρομερή κατάσταση και είναι τώρα σε δεύτερη-τρίτη χρονιά ανάπτυξης. Και το τρίτον, ασχολείστε με το ε, εκπεφρασμένο χρέος των κρατών, το διαπιστωμένο. Αλλά υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος στο έμεσο ε, χρέος των κρατών. Πολλά κράτη-μέλη, ένα είναι και το δικό μου, η Γερμανία, σε ένα-δύο χρόνια θα έχουν σημαντικές δυσχέρειες αν αυτό το έμεσο χρέος, δηλαδή το κόστος των ε, συντάξεων κτλ. δεν ληφθεί υπόψη. Σας ρωτάω λοιπόν, πότε θα αντιμετωπίσετε και αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Κλίνς για τις ερωτήσεις σας. Όσον αφορά την ενιαία αγορά και την καλύτερη ρύθμιση, συμφωνώ μαζί σας ότι δεν μπορούμε να λύσουμε τα οικονομικά προβλήματα της Ευρώπης επικεντρωνόμενοι μόνο στην μακροοικονομική πολιτική. Πρέπει να κοιτάξουμε και άλλα μακροοικονομικά στοιχεία, για παράδειγμα πώς να βελτιώσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον για να έχουμε περισσότερες επιχειρήσεις στην Ευρώπη δημιουργικές και να έχουμε περισσότερες επιχειρήσεις που να μπορούν και να θέλουν να αναπτυχθούν και να βρίσκονται στην Ευρώπη σε καλή κατάσταση. Το κύριο πρόβλημα τώρα, όσον αφορά την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξή της στην Ευρώπη, είναι ότι έχουμε πολλές επιχειρήσεις οι οποίες κάποια στιγμή η ανάπτυξή τους δεν προχωράει όπως στις Ηνωμένε Πολιτείες. Γι' αυτό έχουμε και μικρότερη οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Είναι ένας τουλάχιστον παράγοντας. Όσον αφορά την ενιαία αγορά λοιπόν, ο συνάδελφός μου, ο κύριος Μπαρνιέ, παρουσίασε την πράξη ενιαίας αγοράς προσπαθώντας να συμπληρώσει την ενιαία αγορά, να την ολοκληρώσει. Όσον αφορά τον τομέα των υπηρεσιών, όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας, εξακολουθούμε να έχουμε τεράστιο δυναμικό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε για να προχωρήσουμε περισσότερο με την ενιαία αγορά μας. Το δεύτερο στο οποίο αναφερθήκατε είναι μάλλον σχόλιο σχετικά με αυτά που είπε η κυρία Φερέιρα. Βρίσκω πως είναι πολύ σημαντικό τα κράτη να ενστερνίζονται τα προγράμματα. Υπάρχουν χώρες όπου υπάρχει μεγάλη εθνική ενότητα και αποφασιστικότητα και οι χώρες αυτές έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τις προκλήσεις νωρίτερα ή αργότερα, όπως η Ιρλανδία για παράδειγμα. Είναι πολύ βασικά τα μέτρα που πήραν με αποφασιστικότητα και έτσι να ε, βρεθούν σήμερα σε κατάσταση ανάκαμψης και όσον αφορά την απασχόληση. Για το τελευταίο τώρα που είπατε, Ίσως δεν σας κατάλαβα καλά. Αναφερθήκατε στην τάση του δημοσίου χρέους. Μπορείτε να επανελάβετε, παρακαλώ. Το έμεσο χρέος. Σε πολλές χώρες, μέλη, υπάρχουν τέτοιες προκλήσεις στα συστήματα τα συνταξιδοτικά. Και αυτό αποτελεί μέρος συστάσεων για τις διαδικασίες μακροοικονομικών αποτελεί μέρος δηλαδή και αυτό των μεταρρυθμίσεων που θέλουμε να προωθήσουμε. Που έχει να κάνει και με το προσδόκιμο ζωής. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό για την μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών των χωρών 19 χώρες μέλη από τα 27 μετά την κρίση αποφάσισαν να εφερμόσουν τέτοιες μεταρρυθμίσεις. Είναι ένας πολύ σημαντικός ο τομέας που συχνά περνάει απαρατήρητος και ανοίγει το δρόμο για την βιωσιμότητα των δημοσιονομικών. Τον επόμενο χρόνο έχουμε και το EC 2010 για να συζητήσουμε τι συμβαίνει και σε αυτό το πλαίσιο. Και σίγουρα πρέπει να έχουμε περισσότερο φως σε όλα αυτά τα θέματα των υποχρεώσεων. Από το ECR τώρα. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας. Όπως είπατε, ο δημοσιονομικός τομέας πλήττεται σε πολλά κράτη ο χρηματοπιστωτικό τομέα με συγχωρείτε, πλήττεται σε πολλέ χώρε και αυτό αφορά και τον δίκτυ επισφαλιών. Και σύμφωνα ε, με την τρέχουσα έκθεση που βλέπουμε στις Financial Times και αλλού, βλέπουμε ότι θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι απόψεις σας σε σχέση με τους βραχυπρόθεσμους και ε, μεσοπρόθεσμους στόχους. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε κατά πόσο αυτός ο δείκτης θα ήταν χρήσιμος ως προειδοποίηση για τις εξελίξεις που είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Ναι. That's uh, Σε σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, με το δίκτυ για το χρηματοπιστωτικό τομέα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι προσθέσαμε, μπορέσαμε να προσθέσουμε ένα δίκτυ σε αυτό το βαθμολόγιο. Αν δείτε το ESRB σε σχέση με το επίπεδο επισφάλειας, αυτό είναι ένα σημείο αναφοράς για τον δίκτυ αυτής της επισφάλειας προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα βραχυπρόθεσμο δίκτυ επισφαλιών όπως έγινε από τον Οργανισμό Συστημικού Κινδύνου έτσι ώστε να έχουμε αυτόν τον δείκτη του χρηματοπιστωτικού τομέα σε σχέση με την διαθεσιμότητα και των στοιχείων, έτσι ώστε να μην έχουμε και ρυθμιστικές επικαλύψεις. Γι' αυτό ο βραχυπρόθεσμος ε, δείκτης ε, επισφάλειας που όρισε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συστημικού Κινδύνου είναι ένας αρκετά σημαντικός δείκτης. Αν δείτε λοιπόν την τρέχουσα κατάσταση, Τον τραπεζικό τομέα σχετίζεται με τους απαράβατους όρους για να φτάσουμε στην ανάκαμψη στην καλύτερη και στην καλύτερη απασχολησιμότητα με βάση τους ε, στενούς, αυστηρούς δημοσιονομικούς όρους για την ανάκαμψη και για την, ανάκαμψη, και για την ανάπτυξη, ιδιαίτερα στο νότο της Ευρώπης. Γι' αυτό και η παγίδα ρευστότητας είναι μια δημοσιονομική παγίδα, γιατί τα στοιχεία αυτά σχετίζονται και με τα απαγορευτικά επιτόκια. Τώρα, τι πρέπει να γίνει κατεπηγόντως. Θα πρέπει να δράσουμε και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Η ΕΤΕ πληρεί τα χάσματα εκεί όπου οι ιδιωτικές τράπεζες δεν μπορούν να υποστηρίξουν την πραγματική οικονομία. Η κεφαλαιοχική ε, αύξηση κατά 10 δις ευρώ που αποφασίστηκε επιτρέπει στην ΕΤΕ να δανειοδοτεί φέτος κατά 40%. Η ΕΤΕ βασίζεται και στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή τις ιδιωτικές τράπεζες και τους ε, κεφαλαιοχικούς επενδυτές και πιστεύουμε ότι θα ξεκλειδώσει 180 δις από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για το, την επόμενη τρετία αρχίζοντας από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε την ιδιωτική επένδυση και εδώ δεν μιλάμε για διάσωση των τραπεζών αλλά για ροή πιστώσεων για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Γι' αυτό καλωσορίζω τη δανειοδότηση προς τις ΜΜΕ που ενέκρινε η ΕΤΕ εχθές μέσα στα πλαίσια του, της εντολής δανειοδοτήσεων και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει και σωστή τιτλοποίηση ε, χρεογράφων για τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να υπάρχει ροή κεφαλαίων. Πιστεύω ότι εκτός από την ΕΤΕ θα υπάρξουν και άλλες δυνατότητες επίλυσης του ζητήματος, γιατί είναι μια μεγάλη στενοπός αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει η Ευρώπη για την ανάπτυξή της. Λάμπερτ, εκ μέρους των Πρασίνων τώρα. Ευχαριστώ και καλημέρα, κύριε Επίτροπε. Καλώς ήρθατε. Εμείς οι πράσινοι δεν είμαστε υπέρ των χρεών, τα μισούμε. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει συνταγματική υποχρέωση για τους πολιτικούς της χώρες μέλη να μειώνουν το βάρος το οποίο μεταφέρεται στις επόμενες γενιές. Όλα τα βάρη, όχι μόνο ένα μέρος. Ξέρω ότι εσείς δεν συμμερίζεστε και τέλος πάντων η Γενική Διεύθυνση ΦΥΝ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι άλλοι φίλοι σας υπουργοί στο ΕΚΟΦΗΝ δεν συμφωνούν με αυτήν την ιδέα. Εκεί είναι που διαφέρουμε περισσότερο ιδεολογικά. Δεν μου αρέσουν οι λύσεις ε, που προωθούνται. Θα μπορούσα να τις δεχτώ, εάν όμως υπήρχαν και αποτελέσματα. Αν έβλεπα δηλαδή ότι το δημόσιο χρέος μειωνόταν, τότε θα έλεγα, εντάξει, μπορεί να μην μου αρέσει η συνταγή, αλλά αν μη τι άλλο, δουλεύει. Έχει αποτελέσματα. Αλλά δεν φέρνει αποτελέσματα αυτή η παλιά, η παραδοσιακή συνταγή. Πόσο πρέπει να περιμένουμε ακόμα και τι. Γιατί δεν λειτουργεί. Γιατί δεν εφαρμόζουμε αρκετά καλά τη συνταγή. Γιατί δεν την εφαρμόζουμε αρκετό χρόνο. Πρέπει να περιμένουμε κι άλλο. Τι φταίει που δεν έχουμε επιτυχία. Εγώ αυτό που βλέπω είναι τεράστια ένδια. Οπότε και η ένδια είναι ένα στοιχείο βέβαια του δημοσίου χρέους. Μία μόνο μορφή του. Πολλοί από εσά βέβαια μπορεί να σκέφτονται ότι υπάρχουν πιο θετικά μέτρα. Ανταγωνιστικότητα, σύγκληση, τέτοιου είδου μέτρα. Εσείς πώς βλέπετε αυτά τα μέτρα, ποια νομική βάση θα έχουν, πότε θα έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση και τι εναλλακτικέ λύσεις θα έχουμε επιτάπητος. Δεν ξέρω βέβαια αν θα βοηθήσουν. Να ξέρετε ότι έχω χάσει μεγάλο μέρος της εμπιστοσύνης μου, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Ξέρω ότι εσείς προσωπικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι Υπουργοί Οικονομικών είναι έξυπνοι άνθρωποι ο καθένας, αλλά συλλογικά νομίζω ότι δεν βλέπουν, εθελοτυφλούν. Μήπως θα έχουμε ένα βαθμολόγιο για την επόμενη χρονιά και αν ναι, πείτε το μας και να ξέρουμε και πότε θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε αυτό μαζί σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λάμπερτς. Θα αρχίσω με το τελευταίο που με ρωτήσατε. κατά πόσο θα αλλάξουμε τους δείκτες. Εφόσον το κάνουμε, να ξέρετε ότι πρώτα θα ζητήσουμε την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να προχωρήσουμε βάσει υπεσυμφωνημένης απόφασης. Θα γίνουν δηλαδή διαβουλεύσεις έγκαιρα. Δεν το κάναμε μέχρι τώρα, αλλά θα το διορθώσουμε, να ξέρετε. Και αν χρειάζονται αλλαγέ για το βαθμολόγιο, θα γίνουν. Τώρα, το δεύτερο εξάμεινο της χρονιάς αυτής θα συζητήσουμε και για να αξιολογήσουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο συνολικά. Και θα συζητήσουμε και κατά πόσο το βαθμιολόγιο και οι δείκτες που χρησιμοποιούμε βοηθούν για να μειωθούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Τώρα για την ερώτησή σας όσον αφορά το δημόσιο χρέος. Θέλω εδώ να υπογραμμίσω ότι δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στο δημόσιο χρέος, επικεντρωνόμαστε και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό χρέος. Οι μακροοικονομικές ανισορροπίες και οι σχετικές διαδικασίες αφορούν και τα δύο. Και πολλές χώρες που ελέγχονται με τις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις, Γίνεται αυτό εξαιτία των ανησυχών που υπάρχουν όσον αφορά τις εξωτερικές υποχρεώσεις. Κατόπιν τούτων, Δεν θέλουμε να εξετάζουμε μόνο το δημόσιο χρέος. Κάτι που κάναμε. Έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης επικεντρώνεται στο δημόσιο χρέος και στο έλλειμμα. Και αυτές είναι οι συστάσεις που κάνουμε στις κυβερνήσεις των χωρών μελών. Είναι κατανοητό γιατί Περισσότερα έχουμε να πούμε για τις δράσεις των κυβερνήσεων που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι μπορούμε να πούμε στον ιδιωτικό τομέα. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξετάσουμε και το ιδιωτικό χρέος, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στις χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Και επανέρχομαι τώρα στο μέσο σύγκλησης. Αργότερα σε επόμενες ε, απαντήσεις που θα δώσω γιατί πέρασε ο χρόνος μου. Πρόεδρος. Άκουσα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το web streaming μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκτός Κοινοβουλίου λειτουργούν. Μέσα στο Κοινοβούλιο φαίνεται υπάρχει πρόβλημα με την αναμετάδοση αυτή. Ο Νίκολας Χουντής τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Ρεν, κύριε Αντιπρόεδρε, όλα αυτά τα χρόνια ως εκπρόσωπος της ομάδας της Αριστεράς και ως Έλληνας Ευρωβουλευτής γνωρίζετε ότι σε αυτούς τους διαλόγους στο πλαίσιο των, της Επιτροπής μας, στην Ολομέλεια, στο γραπτό και στον προφορικό έλεγχο, έχουμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας για τις πολιτικές της Κομισιόν, τις αντιρρήσεις μας για τα μνημόνια, την Τρόικα. Δεν θα τα επαναλάβω σήμερα, σας είναι γνωστά. Άλλωστε αρκετοί συνάδελφοι ε, σήμερα στις τοποθετήσεις, σας, συγγνώμη, σας έκαναν κριτική και, ε, σε συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχουν όμως ορισμένα θέματα, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Ρεν, ανεξήγητης και παράξενης συμπεριφοράς της Κομισιόν. Αγαπητοί συνάδελφοι, το τελευταίο παράδειγμα πάνω στο οποίο θέλω να μου δώσει κάποιες διευκρινήσεις ο κύριος Επίτροπος. Στην Ελλάδα, μέχρι πρόσφατα, προωθεί το η συγχώνευση της μεγαλύτερης τράπεζας της Εθνικής με τη Eurobank. Αυτή η συγχώνευση θεωρείται τελειωμένη υπόθεση ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής είχε πει ότι για αυτή τη συγχώνευση έχουμε την έγκριση θεσμικών παραγόντων της Ελλάδας, τη συνένεση της Κομισιόν. Ξαφνικά η Τρόικα και επομένως και η Κομισιόν αλλάζει στάση και λέει να σταματήσει η διαδικασία συγχώνευσης, να γίνει ξεχωριστή η διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στην εθνική ξεχωριστά στη Eurobank και όπως αντιλαμβανόσαστε αυτό γίνεται δύσκολο, όπως αποδείχθηκε και στην πράξη, με συνέπεια να έχουμε την υποχρεωτική μέσω του δημοσίου πέρασμα αυτών των τραπεζών στους ιδιώτες. Αναρωτιέμαι, κύριε Ρεν, τελικά τι έπαθε ο εκπρόσωπός σας, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν στην Τρόικα και κάτι που φαινόταν ότι είχε συμφωνηθεί να το ακυρώνει. Δεν ξέρω αν στη συνέχεια διαπίστωση προβλήματα ανταγωνισμού δεν θα ήταν σοβαρή, κατά τη γνώμη μου, εξήγηση. Αυτό που διαρρέει στα μέσα μαζική ενημέρωση είναι, από την δική σας την πλευρά έτσι λέγεται, είναι ότι αν γινόταν η συγχώνευση θα υπήρχε δυσκολία στη συνέχεια λόγω του όγκου του νέου οργανισμού για την ε, πώλησή του. Αν είναι αυτό, τότε επιβεβαιώνονται όλα αυτά που γράφονται και ενδεχομένω κυκλοφορούν στην Ευρώπη ότι ακυρώθηκε η συγχώνευση με την πρόθεση να απολυθεί η μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα η εθνική έναντι ευτελού ε, ε Το ερώτημα λοιπόν. Τα ερωτήματα τα ανακεφαλαιώνω. Γνωρίζετε κύριε Ρεν αν υπάρχει ενδιαφέρον από κάποια γερμανική τράπεζα για να αγοράσει την εθνική. Δεύτερο, γιατί άλλαξε στάση η Τρόικα, ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν, για μια υπόθεση που φαινόταν ότι είχε συμφωνηθεί. Και πότε θα τελειώσει αυτό το ξεπούλημα τη ελληνική οικονομία. Ευχαριστώ κύριε Χούντι για την ερώτησή σας. Η Ελλάδα δεν είναι τμήμα της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών για τον προφανή λόγο ότι είναι χώρα που υπάγεται στο πρόγραμμα. Η συζήτηση αφορά τις μακροοικονομικές ανισορροπίες με βάση των 13 εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων. Θέσατε την ερώτηση των συγχωνεύσεων τραπεζών και της ανακεφαλαιοποίησης του ελληνικού τραπεζικού τομέα. Θέλω μόνο να πω ότι η Επιτροπή στηρίζει τη διαδικασία αναδιάρθρωσης και ανακεφαλαιοποίησης δίδοντας ε, αποθεματική χρηματοδότηση από τις ε, χώρες μέλη της Ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά δεν είμαι σε θέση να υπησέλθω σε λεπτομέρειες για συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις για την ΑΕΒ τράπεζα. Ε, δεν θα ήταν ε, σκόπιμο κάτι τέτοιο. Το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης βαδίζει ε, με το σωστό ρυθμό και είναι ζωτικό μαζί με τους Έλληνες εταίρους μας, δηλαδή συγκεκριμένα τις ελληνικές αρχές, την ελληνική κυβέρνηση, να επιτύχει η ολοκλήρωση της διαδικασίας διόρθωσης και ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών στην Ελλάδα αποκατάστασης και ανακεφαλαιοποίησης. Είναι ουσιώδης προϋπόθεση για να επανέλθουμε σε βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στη χώρα. αν είναι πιστική η απάντηση προφανώ το ότι η ερώτηση ενδεχομένω είναι εκτό θέματος. Κύριε Επίτροπε πιστεύω ότι είναι εντό του θέματος τουλάχιστον στο σκέλος παρακολούθησα την εισήγησή σα, που λέτε ότι βρισκόμαστε στην παγίδα τη ρευστότητα και υπάρχει ένα φαύλο κύκλο, αν το κατάλαβα καλά. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα των τραπεζών νομίζω υπάρχει αυτό. Αυτό που θέλω να σα πω και τελειώνω, ναι, τελειώνω, τελειώνω, ότι αυτή η παρατήρηση, αυτό το ερώτημα, που είναι άκρο πολιτικό, όπω είπατε στην αρχή πω πρέπει να μιλήσουμε, δεν εκφωνείται μόνο από μένα που σα είπα ότι έχουμε μια ε, ριζική αντίρρηση. Εκφωνείται από κορυφαίου, όπω τα ξέρετε, πολιτιακού παράγοντε τη δημοκρατία τη Ελλάδα. Και επομένω χρειάζεται πιστική απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να τη δώσετε. Um, δεν υπάρχει χρόνος για να απαντηθεί στην πλωματική ερώτηση. Υπάρχουν θέματα τα οποία δεν απαντήθηκαν και ε, με βάση αυτά που ήδη υπόθηκαν για το αν υπάρχει έλλειψη κατανόησης ε, όσον αφορά κάποιες αποφάσεις της Τρόικας, πρέπει κάπου να υπάρχει ένας μηχανισμός ούτως ώστε να λάβουν απαντήσεις. Ε, αν μπορείτε να μας πείτε τίποτα περισσότερα στη συνέχεια γραπτός, θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα. Ή θα πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα αυτό όταν θα έχουμε προσώπους της Τρόικα παρόντες. Ε, από το EFD, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι για την παρουσία σας, ε, κύριε Επίτροπε. Ας επανέλθουμε σε θέματα δημοσιονομικής πειθαρχίας. Από την αρχή της δημοσιονομικής ε, κρίσης μας είπατε ότι αν υπάρχουν αυστηροί κανόνες θα μπορέσουμε να απαλύνουμε την κρίση και τις υπερβολικές ε, μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ακολουθήσαμε τους ε, κανόνες και πριν από την κρίση είχαμε το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας, αλλά δεν ακολουθήθηκε πάντα σωστά από όλους. Θεωρούσαμε ότι πρέπει να υπάρχει δημοσιονομική πειθαρχία παράλληλα με μέτρα λιτότητας. Στο μεταξύ αλλάξατε άρδιν. Δώσατε εξαιρέσεις σε κράτη-μέλη ως προς τα μέτρα λιτότητας και επεκτείνετε το πεδίο σας. Με τις εξαιρέσεις αυτές τα μέλη της Ευρωζώνης μπορούν να ακολουθήσουν την παλαιά ανισόρροπη δημοσιονομική τους πολιτική. Άρα, αρχικά, ορισμένες χώρες δεν ακολούθησαν το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τώρα τους χορηγείται και εξαιρέσει σε σχέση με τους αυστηρούς κανόνες. Δηλαδή, δεν ακολουθούσαμε τους κανόνες πριν, δεν τους ακολουθούμε και τώρα. Άρα κύριε Επίτροπε, με όλη αυτή τη νέα νομοθεσία και με τις συνθήκες, ποια είναι η ουσία αν δεν ακολουθούμε και τους νέους κανόνες. Τι έχουμε επιτύχει πέρα από την περισσότερη ρύθμιση και μεγαλύτερο διοικητικό φόρτο. Απάντηση. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Σε σχέση με τα προλεγόμενα της ερώτησής σας, η αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης είχε ένα διτό αποτέλεσμα. Εστιάσαμε την προσοχή μας ε, στην διαρθρωτική βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών και δεν σταθήκαμε τόσο σε ονομαστικούς στόχους. Και αυτό για να ανταποκριθούμε στα λεγόμενα πρώην ενός πρώην επιτρόπου που είπε ότι το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης είναι γελίο υπάρχουν περισσότερα περιθώρια ελιγμών και μπορούμε να σταθούμε στην διαρθρωτική βιωσιμότητα και όχι σε ονομαστικούς στόχους. Γι' αυτό το ε, σύμφωνο σταθερότητας έγινε και πιο σοβαρό, αντιμετωπίζοντας και τους κύκλους συστημικού κινδύνου. Οι νέοι κανόνες επίσης προβλέπουν ένα μηχανισμό ενίσχυσης και αυτό το είδαμε έμπρακτα. Τα κράτη-μέλη λοιπόν λαμβάνουν υπόψη πιο σοβαρά τους κανόνες, διαφορετικά θα υποστούν δημοσιονομικές κυρώσεις. Άρα, βράχει και μέσο πρόθεσμα, καθώς και μακροπρόθεσμα, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα βοηθήσει για να ε, μπορέσει να αποτρέψει κρίσεις όπως αυτή που ζήσαμε πρόσφατα. Παράλληλα όμως υπάρχει και αυτή η μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης, μεταρρύθμιση και αναθεώρηση αυτών των κανόνων, έτσι ώστε να προλάβουμε και να ανταποκριθούμε στους στόχους μας. Ως προς τις εξαιρέσεις τις οποίες ε, προαναφερθήκατε, σε σχέση με τις ε, προθεσμίες για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος, λάβαμε υπόψη τη διαρθρωτική δημοσιονομική προσπάθεια που ε, προέβαλαν αυτές οι χώρες με βάση και το γενικό τους outlook. Έτσι, μπορούν να γίνουν διορθώσεις του υπερβολικού ελλείμματος όπως έγινε πέρσι με την Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα. Ίσως να ισχύσει φέτος την Άνοιξη και για ορισμένες άλλες χώρες αν πληρούνται οι όροι. Αλλά είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας για την ίδια τη χώρα, για το λαό της και για τους υπεύθυνους πολιτικούς της. Μιλάμε λοιπόν για ανάλογο ρυθμό προσαρμογής. Και εδώ αναφέρομαι στην Ιρλανδία και τη Λετωνία, οι οποίες έλαβαν τάχιστες αποφασιστικές δράσεις και έτσι μπορούν να έχουν ανάκαμψη και καλύτερη απασχόληση. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους του ΕΛΚ τώρα, η Κορίν Βόρτμαν Κόλ. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε, που είσαστε εδώ σήμερα είπατε για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης. Θέλω να σας ενθαρρύνω να χρησιμοποιήσετε τις νέες σας εξουσίες με έναν δίκαιο και ανεξάρτητο τρόπο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύ πολιτικό λόμπι από διάφορες χώρες, μικρές και μεγάλες, αλλά είναι σημαντικό εσείς να χρησιμοποιήσετε τις εξουσίες που έχετε με σαφήνεια. Αναφερθήκατε στους δείκτες. Ναι, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει χαμηλή ανάπτυξη, υπάρχει και δυσκολία των χωρών να συλλέξουν τους φόρους. Και γι' αυτό ίσως και ο δρόμος προς τις δευτερωτικές μεταρρυθμίσεις είναι τόσο αργός. Τα είπαμε χτες και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τώρα εγώ θέλω να μου μιλήσετε λιγάκι για τον οικονομικό κύκλο και το πακέτο των 6 ο πρόεδρος Μπαρόσο και στις ΗΠΑ Πολιτείες αλλά και όπως το μετέφεραν τα μέσα ενημέρωσης στην Ευρώπη αναφέρθηκε ουσιαστικά σε μια πιο ήπια εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών και των μεταρρυθμίσεων ακριβώς επειδή υπάρχει λιτότητα. Μερικές φορές πρέπει κανείς να πάρει κάποια μέτρα βραχυπρόθεσμα σκληρά για να μπορέσει αργότερα να εποφεληθεί η απασχόληση. Τα κράτη-μέλη λοιπόν τα οποία έχουν παρουσιάσει τα προγράμματά τους για τις διαδικασίες υπερβολικών ελλημάτων και είναι πάνω από το μείον 3 για το 2014, θα επεκταθούν οι προθεσμίες για αυτές τις χώρες. Και όταν δεν έχουν συγκεκριμένα μέτρα όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Επειδή όταν τα κράτη-μέλη παρουσιάζουν μια ωραία υπόσχεση ότι θα τηρήσουν τα κριτήρια για τα επόμενα χρόνια, αλλά τελικά δεν τα καταφέρνουν. Εσείς θα δέχεστε τέτοια προγράμματα ως έχουν. Ευχαριστώ. Τρία πράγματα θέλω να σας πω. Πρώτον, αυτό που λέτε εσείς lobbying εγώ το λέω εταιρική σχέση, συνεργασία, που είναι στην καρδιά των μεταρρυθμίσεων και της οικονομικής διακυβέρνησης. Νομίζω ότι έχουμε επικοδομητικό διάλογο με όλες τις χώρες μέλη. Προσπαθούμε μαζί να βρούμε λύσεις όχι μόνο μέσω της οικονομικής εξυγίασης, αλλά και μέσω των διορθωτικών μεταρρυθμίσεων. Γιατί επηρεάζουν την ανάπτυξη και τα δημοσιονομικά και πρόθεσμα και όχι μόνο βραχυπρόθεσμα όπως γίνεται με τις, ε, τη δημοσιονομική εξυγένση. Τώρα, η δημοσιονομική εξυγένση κατά πόσο βασίζεται υπερβολικά στους φόρους και ότι έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη. Όπως είπατε, σε πολλές χώρες μέλη, δυστυχώς, η άσκηση αυτή της δημοσιονομικής εξυγίανσης βασίστηκε πάρα πολύ στην αύξηση των φόρων αντί για την μείωση των δαπανών. Είναι μεγάλη δυσκολία πολιτικά, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο θετικός αντίκτυπος στην ανάπτυξη. Τρίτον, όσον αφορά τη γενική προσέγγιση. Όχι, δεν υπάρχει γενικευμένη παράταση των προθεσμιών και αυτό για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί οικονομικά δεν θα έχει νόημα. Υπάρχουν πολλές χώρες που και μπορούν και θέλουν να μειώσουν φέτος τα υπερβολικά του ελλείμματα και εμείς αυτό θέλουμε να το στηρίξουμε. Δεύτερον, δεν ευθυγραμμίζεται κάτι τέτοιο με το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Είναι προτιμότερο, πιστεύω, να έχουμε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση βάσει του συμφώνου αυτού, ώστε να δούμε τις προκλήσεις, τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία σε κάθε χώρα μέλη και ανάλογα να προσαρμόσουμε την πολιτική μας και οι χώρες να τηρούν το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης παρά να παίρνουν από μόνες τους τις αποφάσεις τους. σε ευχαριστώ. Ο Γιώργο Θέο τώρα, εκ μέρους του, ε, του ΕΛΚ επίσης. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Σε μια απάντηση που δώσατε ε, λίγο, λίγη ώρα πριν στην Ελίζα Φερέιρα, είπατε ότι η Πορτογαλία εδώ και δύο χρόνια βρισκόταν σε μια κατάσταση μη βιώσιμη, γιατί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Είναι γεγονός ότι επρόκειτο για εθνική πολιτική ανευθυνότητα για μερικά χρόνια. Γι' αυτό μπήκαμε κι εμείς υπό πρόγραμμα προσαρμογής το οποίο αξιολογεί, η Τρόικα σε τακτά χρονικά διαστήματα και το αποτέλεσμα είναι θετικό. Όπως θα γνωρίζετε, είναι πολύ δύσκολο να αυξηθούν οι εξαγωγές. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Ο μεγαλύτερος μας εταίρος, η Ισπανία, γνωρίζει συρρυκνούμενη επίσης οικονομία, όπως είναι και η δική μας. Η ανεργία έχει αυξηθεί σε μη βιώσιμα επίπεδα. Η κοινωνική και πολιτική συνένεση είναι αξιοθρύνητη δεν θεωρείτε ότι η Πορτογαλία χρειάζεται περισσότερα κίνητρα. Έγινε λόγος για ληξιπρόθεσμους τίτλους, για ε, προέκταση του περιθωρίου προσαρμογής. Δεν θα ήταν σκόπιμο αυτή η προσαρμογή να προσαρτάται σε μία αναπτυξιακή πολιτική γιατί μιλάμε για το καρότο και το μαστίγιο. Πολλά μαστίγια είδαμε και πολύ λίγα καρότα. Η Ελίζα Φερέιρα είπα «Φτάνει πια». Εγώ θέλω να σας πω να μας προβάλλετε μία εναλλακτική λύση, αναπτυξιακής μορφής. Έτσι ώστε να απαλληφθούν τα μαστίγια και να έχουμε περισσότερα καρότα υπομορφή κινήτρων. Μπορούμε να πιστεύουμε σε κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όπως απάντησα και στον κύριο Χουντή, απαντώ και σε εσάς. Η Πορτογαλία δεν εντάσσεται στο, στη διαδικασία μακροοικονομικών ισορροπιών γιατί είναι χώρα υποπρόγραμμα προσαρμογής. Εφόσον όμως με ρωτήσατε, θα σας δώσω μία απάντηση όσο καλύτερα μπορώ. Λάβαμε αποφάσεις για να υποστηρίξουμε την οικονομική προσαρμογή της Πορτογαλίας ουσιοδός. Πρόσφατα Δύο εβδομάδες πριν θα θυμόσαστε ότι το Eurogroup με την υποστήριξη της Επιτροπής έλαβε αποφάσεις για την Ιρλανδία και την Πορτογαλία σε σχέση με τους ληξιπρόθεσμους, με τα ληξιπρόθεσμα δάνεια. Μέσα στα πλαίσια της χρηματοδότησης της αγοράς και της εξόδου από το πρόγραμμα. Η Ιρλανδία βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία, αλλά πιστεύω ότι και η Πορτογαλία θα είναι επιτυχής και θα μπορέσει να εξέλθει από το πρόγραμμα και να χρηματοδοτήσει την αγορά της, να ξαναμπεί στις αγορές. Αυτός είναι και ο στόχος που συμμεριζόμαστε όλοι σε αυτή την αίθουσα. Να μην έχουμε δηλαδή προέκταση του προγράμματος, αλλά να εξέλθετε από το πρόγραμμα και να ξαναμπείτε στις αγορές, όπως είπε και στην κυρία Φερέιρα. Γι' αυτό ακριβώς ε, μιλήσαμε και για την παράταση της λήξης ομολόγων, των ομολόγων. θα λάβουμε υπόψη αυτή την ε, προέκταση, την παράταση και φέτος, διότι το οικονομικό outlook ήταν λίγο χειρότερο από το αναμενόμενο. Οι χώρες πρόγραμμα θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτή την οδό εμπρόθεσμα και προβλέπεται και μια διαδικασία επισκόπησης λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία τα οποία είναι λίγο χειρότερα από ότι τα αναμενόμενα. Γι' αυτό η διαδικασία μεταρρυθμίσεων συνεχίζεται στην Πορτογαλία και μαζί με τους Πορτογάλους συναδέλφους προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στη δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση στη Νότιο Ευρώπη, διότι ιδιαίτερα στην Πορτογαλία οι συνθήκες δανειοδότησης είναι δυσμενείς και δημιουργούν μια μεγάλη στενοπό για την αντιμετώπιση των ζητημάτων μας. Πρόεδρος, θα πρέπει να επιταχύνουμε. Ε, τώρα ε, ο κύριος Μπόρμαν από τους Σοσιαλιστές. Κύριε Επίτροπε, καίγεται η Ευρώπη, κύριε Επίτροπε. Η κατάσταση δεν είναι τόσο ευχάριστη ως εδώ. Η ανεργία των νέων εκρήγνεται, τα χρέη εκρήγνεται, ιδιαίτερα εκεί όπου δρά η Τρόικα και καταραίει η ανάπτυξη. Πρέπει να διευκρινίσουμε συγκεκριμένα ερώτημα, ερωτήματα. Έχει αρκετό νερό η πυροσβεστική υπηρεσία θα σβήσει τις πυρκαγιές ή θα μιλάει για ε, να σβήνουν οι πυρκαγιές που θα συνεχίσουν να καίνε. Τι έγινε το σύμφωνο ανάπτυξης που θέλαμε να αντιμετωπίσουμε τις ανισορροπίες μέσω αυτού στο οποίο ε, είχαν αποδοθεί 120 δις και εμείς ε, θεωρήσαμε ότι είναι ανεπαρκή. Δεν είναι το μεγάλο ψέμα. Πού είναι αυτά τα 55-60 δις που θα έπρεπε να ε, ξοδευτούν στοχευμένα από ευρωπαϊκούς πόρους η εγγύηση για τους νέους, 6 δις, πολύ μικρή, περιεκόπη. Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας μας λέει ότι χρειάζονται 100 δις, 100 δις πρέπει να δοθούν όχι για να καταπολεμήσουμε απλώς την ε, ανεργία των νέων, αλλά για να ε, δώσουμε τα αναγκαία επιδόματα για να μπορέσουν να επιζήσουν οι νέοι. Θα αυξήσετε, παρακαλώ, τις πιστώσεις. Πόσα, πόσες πιστώσεις ούτως ή μέχρι στιγμής δεν αξιοποιούνται γιατί δεν μπορούν να δώσουν τη συμπληρωματική χρηματοδότηση στα κράτη-μέλη. Πώ θα καταπολεμήσουμε την ανεργία, πώ θα βοηθήσουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Έχετε ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει συζητήσει για αυτό. Το χειρότερο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν πιστεύουν πια οι άνθρωποι ότι μπορεί να αλλάξει κάτι πολιτική. Πρέπει να σταματήσουμε να μην έχει πρόσωπο κάνει η Τρόικα. Ποια είναι αυτή η Τρόικα. Αν θέλουμε να του τηλεφωνήσουμε, δεν έχουμε πού να του τηλεφωνήσουμε. Δεν έρχονται στα κοινοβούλια, δεν μιλάνε με εμά οι Τροϊκανοί. Πέστε μας παρακαλώ, ποια είναι η προσωπική σας άποψη. Τα κράτη-μέλη είναι που φταίνε. Ποια κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για αυτή την πολιτική. Να μας πείτε ποια είναι. Για το ότι ασκούμε εντελώς λανθασμένη πολιτική ή όπως πριν φταίει η Γενική Διεύθυνση ΕΚΦΗΝ η οποία κάνει τη μία λανθασμένη πρόγνωση μετά την άλλη. Πότε θα σταματήσουν αυτά τα πράγματα. Πότε θα, αρχίσουμε, θα σταματήσουμε να ε, εργαζόμαστε με τέτοιο ιδεολογικό τρόπο. Πότε θα αρχίσουμε να λαμβάνουμε υπόψη την πραγματική κατάσταση, τα πραγματικά στοιχεία. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Είναι σημαντικό, πιστεύω, να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ και να προωθήσουμε την ε, γενική κοινωνική ατζέντα. Να την εφαρμόσουμε με ευρύ πνεύμα. Στο σχέδιο της Επιτροπής για το συντονισμό, την επιτήρηση και τη στήριξη της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών, όλα αυτά πρέπει να ενισχυθούν στα πλαίσια της διακυβέρνησης της ΟΝΕ, ιδιαίτερα στους τομείς που έχουν άμεση σχέση με τις ε, πολιτικές απασχόλησης και τη λειτουργία της Ευρωζώνης. Ο συνάδελφός μου, επίτροπος που είναι αρμόδιος, ε, θα υποβάλει μία ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της άνοιξης για το θέμα αυτό. Εργάζεται ήδη έντονα για τον τομέα αυτό. Έχουμε εντείνει τις πολιτικές απασχόλησής μας για να παράσχουμε για κάθε νέο στην Ευρώπη μία δυνατότητα είτε εκπαίδευσης, είτε κατάρτισης, είτε μιας θέσης μαθητείας. Αυτός είναι ο στόχος του προγράμματος ε, εγγυήσεων για τους νέους, που βασίζεται στις θετικές εμπειρίες που είχαμε, για παράδειγμα στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπου λειτουργεί ήδη με εδώ και 22-25 χρόνια, αν θυμάμαι σωστά. Και βέβαια δεν υπάρχει καμιά πανάκια, αλλά δίνει στους νέους τη δυνατότητα είτε να βρουν θέση απασχόλησης, είτε εκπαίδευσης, είτε κατάρτισης. Όλα αυτά είναι ουσιώδη για να έχουν μια δυνατότητα να εισέλθουν στην αγορά εργασίας όταν θα βελτιωθεί η κατάσταση στη χώρα τους. Για τη λειτουργία τώρα της Ευρωζώνης και της Τρόικα. Καλωσορίζω αυτό που είπε και η Πρόεδρος και ο κύριος Μπόρμαν να το συζητήσουμε σε περισσότερο βάθος στο μέλλον. Είναι σαφές ότι η δομή της λήψης αποφάσεων και της διακυβέρνησης στα πλαίσια της Τρόικα είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και βαριά. Διότι όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ευρωζώνη στα πλαίσια της Τρόικα λαμβάνονται από 17 κράτη-μέλη ομόφωνα. Συνήθως ε, αυτό χρειάζεται και την θετική συνένεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Γιατί όλοι αυτοί ε, συμβάλλουν οικονομικά στα μέτρα. Η οικονομική συμβολή της Κομισιόν ε, βασίζεται στο μηχανισμό, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ασφάλειας και ε, Σταθερότητας αλλά αυτός ο οργανισμός η e FSM, επειδή υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις, δεν θα χορηγήσει νέα δάνεια στα πλαίσια του ESM, γιατί το ε, μόνιμο ESM θα ε, αρχίσει να λειτουργεί πλήρως. Υπάρχουν 20 ε, κόκκινες γραμμές, 20 σημεία στα οποία μπορεί να ισχύσει βέτο. Άρα είναι πολύ δύσκολο να υπάρξουν ε, συγκεκριμένες αποφάσεις. Και κατά συνέπεια οι αποφάσεις που λαμβάνονται πολλές φορές δεν είναι οι βέλτιστες αλλά οι αμέσως χειρότερες. Είμαι διατεθειμένος να το συζητήσω. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να αξιοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα η κοινοτική μέθοδος. Αυτή θα οδηγούσε σε καλύτερες λύσεις. Πρόεδρος. Υπήρχαν 20 έτσι κι αλλιώ ε, και 20 κόκκινες γραμμές από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκ μέρου του ΕΛΚ, ο Χερμπέρτ Τόφμαν έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Να κάνω μία ερώτηση που την ανέφεραν και κάποιοι προηγούμενοι. Είπαν ότι οι πολίτες ε, δεν αποδέχονται αυτά τα οποία κάνουν. Υπάρχει τέτοιο θέμα. Έρχομαι από την Ιταλία. Μπορεί να μην το περιμένατε επειδή δεν μιλάω Ιταλικά, αλλά εάν εξετάσω την κατάσταση και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες όπως τη Γαλλία, όπου βλέπουμε τι γίνεται και με τις εκλογές, δεν είμαι τόσο αισιόδοξο όπως και εσείς, όσο εσείς για το θέμα συνεργασίας με τα κράτη-μέλη. Διότι διάφοροι ε, βασικοί πολιτικοί και όχι μόνο ευρω, ευρωσκεπτικιστές ε, εκφράζονται διαφορετικά. Γίνονται προεκλογικές εκστρατείες όπου ο εχθρός είναι οι Βρυξέλλες και όπου οι πολιτικοί στην προεκλογική εκστρατεία υπόσχονται ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί θα καταργηθούν εάν αυτοί οι πολιτικοί αναλάβουν την κυβέρνηση. Δεν είναι τόσο λοιπόν ε, ε, αγαστή συνεργασία όσο λέτε. Θα πρέπει λοιπόν να επιχειρήσουμε να αυξήσουμε την αποδοχή από τους πολίτες αυτών που κάνουμε. Προτείνατε ε, να υπάρξει αυτό το μέσο σταθερότητας και σύγκλησης. Από ό,τι κατάλαβα, είναι αυτό που προηγουμένως ο συνάδελφος Φέο αποκάλεσε λουκούμι ή βούρδουλα. Ε, και είπε ότι κυρίως είναι βούρδουλας, δεν υπάρχει αρκετό λουκούμι. Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει περισσότερη αποδοχή στα κράτη-μέλη. Και τι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Γιατί βλέπουμε ότι ορισμένοι αξιοποιούν ε, προεκλογικές εκστρατείες για να καταγγείλουν την Ευρώπη δεν θεωρείτε ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν περισσότερο και τα εθνικά κοινοβούλια και να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη. Γιατί αν δεν το επιτύχουμε αυτό, πιστεύω ότι στο τέλος οι πολίτες δεν θα τα εγκρίνουν όλα αυτά και άρα μακροπρόθεσμα θα αποτύχουμε. Ευχαριστώ. Στις προηγούμενες απαντήσεις μου αναφέρθηκα και θα ήθελα ευρύτερα να συζητήσουμε πώς οι διάφορες χώρες αστερνίζονται τα μέτρα, να το συζητήσουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται πάντα σε επικοδομητικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο όσον αφορά τις πολιτικές που εφαρμόζουμε για την οικονομική και δημοσιονομική μας στρατηγική. Όσον αφορά την αποδοχή από πλευρά λοιπόν των Ευρωπαίων πολιτών, εγώ αντιλαμβάνομαι απόλυτα ότι οι χώρες, πολλές χώρες, έχουν να πάρουν πολύ δύσκολες αποφάσεις, ευάλωτες χώρες. Από την άλλη, δεν είμαι πεπισμένος ότι χωρίς την Ευρώπη ή χωρίς τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οικονομική προσαρμογή θα ήταν πιο εύκολη. Πιστεύω ότι ενωμένοι έχουμε μεγαλύτερη δύναμη. Και γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε την ενιαία μας αγορά, πρέπει να στηρίξουμε τις χώρες μέλη, τις προσπάθειες που κάνουν για μεταρρυθμίσεις και πιστεύω ότι έχουμε πολύ περισσότερα να κερδίσουμε συνεργαζόμενοι μεταξύ μας αντί να προσπαθούμε να επαναθνικοποιούμε ευρωπαϊκές πολιτικές. Όσον αφορά τώρα τη σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα. Το εργαλείο αυτό το οποίο παρουσιάστηκε ε, το Μάρτιο υπάρχουν δύο προτάσεις για τον εκ των προτέρων συντονισμό των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και η άλλη είναι για την ανταγωνιστικότητα. Αυτό σημαίνει ότι τα σχέδια για τις πιο σημαντικές ε, μεταρρυθμίσεις συζητιώνται μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων πριν να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο οι τελικές αποφάσεις. Πιστεύω ότι είναι ένα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη ιδιαίτερα. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, το μέσο συντονισμού και ανταγωνιστικότητας είναι ένα μέσο αλληλεγγύης. Είναι ένα μέσο το οποίο περιλαμβάνει συμφωνίες οι οποίες θα ενισχύσουν ακριβώς αυτό το αίσθημα αποδοχής από πλευράς των Ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Κάποια χώρα μέλη αναλαμβάνει μια δέσμευση για να εφαρμόσει δύσκολες μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τις ενταξιοδοτήσεις, θα μπορούσε να τύχει στήριξη για ένα πρόγραμμα διαβίου κατάρτισης. Αυτά. Τελείωσα. Πρόεδρος, περνάει ο χρόνος. Έχουμε άλλους τέσσερις Προτείνω λοιπόν δύο, να υποβληθούν οι ερωτήσεις και να προσπαθήσουμε όχι δέκα λεπτά για τις δύο αυτές ερωτήσεις, λιγότερο. Ντομινίτσι και Ρόδι μετά. Παρακαλώ. Κύριε Πίτροπε, σε μία συζήτηση και σε ένα λόγο σας τον Απρίλιο στη Monetary and Financial Committee αναφερθήκατε στο χρέος της Ευρωζώνης. 88% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης στα τέλη του 2011 και 93,1% το 2012 και προσδοκία 90,1% 95,1 για το 13. Εσείς απαντώντας στον συνάδελφο Λάμπερτς είπατε ότι λαμβάνετε υπόψη άλλες μεταβλητές και παράγοντες. Όμως είπατε ότι οι πολιτικές σας ε, θέλουν, έχουν σαν στόχο τη συρρήκνωση του υψηλού επίπεδου χρέους, του υπέρογκου χρέους. Μας προτείνετε είναι μία λιτότητα με ανθρώπινο πρόσωπο, γιατί λέτε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε δημοσιονομική εξυγίανση κατά τρόπο φιλικό προς την ανάπτυξη. Στις 9 Απριλίου στο Όσλο όμως, μιλώντας για την Ιταλία, λέτε ότι η Επιτροπή επέτρεψε στην Ιταλική κυβέρνηση να ξεμπλοκάρει το χρέος του δημοσίου έναντι των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση της Ιταλίας κατά τα τελευταία χρόνια. Έτσι πιστεύετε ότι ισχύει ένα φιλικό προς την ανάπτυξη μοντέλο. Η κυρία Κράτσα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θεωρώ πολύ σημαντικό ότι συζητούμε το θέμα των μακροοικονομικών ανισορροπιών καταρχάς, όπως είπε πρόσφατα η κυρία Λαγκάρντ ε, ανισότητα και υγιής ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξουν. εξάλλου ξέρετε το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με κάθε ευκαιρία ε, σημείωσε πόσο είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανισορροπίες για τη σταθερότητα και όχι μόνο της οικονομίας μας αλλά και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού σχεδίου ενοποίησης. Αναφερθήκατε ότι στη μεγάλη, η μεγάλη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα είναι η δημοσιονομική προσαρμογή και οι μεταρρυθμίσεις. Και το κλίμα που υπάρχει σήμερα είναι πολύ ευνοϊκότερο. Αναμφισβήτητα υπάρχει ένα κλίμα σταθερότητας και στρατηγικής, αλλά οι Ευρωπαίοι πολίτες στις ανησυχίες των οποίων αναφέρθηκαν οι συνάδελφοί μου και το ζωέντονα στη χώρα μου την Ελλάδα, θέλουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, όχι μόνο για την προσωπική του ζωή, αλλά και για την βιωσιμότητα της οικονομίας τους και της Ευρώπης. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, οι πολιτικές λιτότητας και δημοσιονομικής προσαρμογής όπως έχουν εφαρμοστεί έχουν αποτελέσματα βιώσιμου κλεισίματος της ανταγωνιστικότητας που είναι το μεγάλο ζητούμενο σήμερα στις ευρωπαϊκές οικονομίες και σας ανησυχεί αυτή η άνοδος του δημοσίου χρέους στις χώρες που υφίστανται αυτό τα προγράμματα. Επίσης ήθελα να σας πω να μας δώσετε μια πιο συγκεκριμένη ε, απάντηση γιατί ήδη ε, απαντήσατε σε επιμέρους ε, θέματα ποια είναι η αλληλοεπίδραση, το συμπέρασμα που έχετε εξάγει από την αλληλοεπίδραση και την αποτελεσματικότητα της λιτότητας αυτή τη στιγμή και των δομικών μεταρρυθμίσεων. Πώς μπορεί να συνεπάρξουν σε μια πορεία βιώσιμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και τις πολιτικές, όχι μόνο τις οικονομικές βέβαια. Σας ευχαριστώ. Και οι δύο ερωτήσεις του κυρίου Ντομίνιτσι και της κυρίας Κράτσα αναφέρονται στο επίπεδο χρέους και το συσχετισμό με την οικονομική ανάπτυξη. Αυτός ο συσχετισμός είναι περίπλοκος και εξαρτάται από κρατικές ιδιαιτερότητες. Δεν υπάρχει ένας ενιαίος κανόνας ή επίπεδο όταν μιλάμε για το δημόσιο χρέος. Και τη στιγμή που είναι ε, ένα σπήλος στην οικονομική ανάπτυξη. Η κοινότητα των οικονομολόγων και όσοι ορίζουν πολιτικές συγκλίνουν σε δύο ζητήματα, σε δύο θέματα. Το υψηλό δημόσιο χρέος έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη. Είτε είναι γραμμικής φύσης, είτε όχι. αποτελεί και τη βάση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σημαίνει ότι το επίπεδο δημοσίου χρέους θα πρέπει να παραμείνει κάτω από το 60%. Επίσης, οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές έχουν βραχυπρόθεσμα επιπτώσεις στη δημοσιονομική εξυγίανση γιατί μιλάμε για μηδενική ανάπτυξη και μέσα στα πλαίσια της νομισματικής μας πολιτικής. Γι' αυτό θα πρέπει να προβούμε σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και σε επενδύσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, διατηρώντας μία πολιτική συνεκτική δημόσιας εξυγίανσης. Όταν μιλάμε για χώρες υποπρόγραμμα, όπως την Ελλάδα, υπάρχει ένας επιπρόσθετος παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη μέσα στα πλαίσια της λήψης πολιτικών αποφάσεων. Είναι οι περιορισμοί και οι όροι του προγράμματος χρηματοδότησης για τις χώρες αυτές. Δηλαδή θα θέλαμε μία πιο συνεκτική δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά αυτό σημαίνει περισσότερη χρηματοδότηση από τις χώρες πιστωτές, το οποίο σημαίνει απόφαση, συναπόφαση του Eurogroup. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία σε σχέση με την οικονομική προσαρμογή στην Ελλάδα ή στην Πορτογαλία. Εάν πιστεύετε ότι η οικονομική προσαρμογή που ισχύει και στη χώρα μου, που όπως είπα ακούω και στη χώρα μου πολλές ανησυχίες, αν θεωρείτε λοιπόν ότι η προσαρμογή αυτή χρειάζεται και επιπρόσθετη απόφαση από το Κοινοβούλιο. Αυτό αφορά τις 14 χώρες πιστωτές της Ευρωζώνης. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ορθολογική πολιτική λήψη αποφάσεων και στην Ευρωζώνη. Πρέπει να προχωρήσουμε, λέει η Πρόεδρος. Γιατί μιλάτε για χώρες πιστωτές και όχι χώρες εγγυήτριες, γιατί δεν χορηγούν χρήματα, εγγυώνται για αυτά και είναι πολύ αρνητικό για τη δημόσια εικόνα μας τη στιγμή που δεν έχουν μεταβεβαστεί χρήματα. Απλώς οι χώρες αυτές είναι εγγυήτριες, χώρες εγγυήτριες και όχι πιστότριες χώρες. Δανειοδοτούν. Τα αγγλικά δεν είναι η μητρική μου γλώσσα. μιλώ για πιστώσεις που καλύπτονται από εγγύησεις. Πρόεδρο, ίσως θα ήταν ε, πιο θετικό εάν μιλάγαμε για εγγυήσει. Η κυρία Ποδηματά και μετά τρεμόζαν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ διπλά για αυτήν την πολύ επικοδομητική ε, παρατήρηση. Ε, μου δίνει αφορμή κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής να σας θέσω το ερώτημα με βάση τις τελευταίες παρατηρήσεις σας απατώντας τους προηγούμενους συναδέλφους αναφερόμενος στις χώρες που εφαρμόζουν ε, πρόγραμμα προσαρμογής είπατε εάν σας κατάλαβα καλά ότι θα προτιμούσατε θα προτιμούσε η ευρωπαϊκή επιτροπή μια πιο ήπια δημοσιονομική προσαρμογή αλλά αυτό θα απαιτούσε ε, περισσότερα χρήματα στα προγράμματα οικονομικής υποστήριξης και άρα αποφάσεις από τα κοινοβούλια των χωρών που δίνουν τις εγγυήσεις στον ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας. Ε, οι συνάδελφοι πριν αναφέρθηκαν στην κατάσταση στην πορτογαλία την κατάσταση στην ελλάδα την ξέρετε είμαστε στην έκτη διαδοχική χρονιά ύφεσης με μια ανεργία που έχει ξεπεράσει το 27%. Οι προβλέψεις λένε ότι φέτος θα, πετύχουμε ένα ε, μηδενικό ε, έλλειμμα δημοσιονομικό και του χρόνου ελπίζουμε να φτάσουμε σε πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα ε, το ερώτημα που θέλω να σας κάνω ε, κύριε αντιπρόεδρε είναι εάν για την περίπτωση της ελλάδας με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα ύφεση τρομακτική ανεργία προτίθεται η ευρωπαϊκή επιτροπή να ενεργοποιήσει και πώς την περίφημη ρήτρα ύφεσης που υπάρχει στο πρόγραμμα. αυτό είναι το ένα ερώτημα. το δεύτερο ερώτημα αφορά την διαφάνεια και τη λογοδοσία σε σχέση με τη λήψη των αποφάσεων τον Τρόικα. Έγινε μεγάλη συζήτηση πριν από τον Ούντο Μπούλμαν, από την κυρία Πρόεδρο. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η συνάδελφός μου η Ελίζα Φερέιρα και εγώ είχαμε προτείνει προς την Επιτροπή προ καιρού να ενταχθούν οι χώρες που εφαρμόζουν πρόγραμμα στη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών εντάσσοντας στοιχεία του προγράμματος προσαρμογής στις συστάσεις αναχώρα διότι αυτό θα βελτιώσει κυρία την πρόεδρε τη διαφάνεια και θα επιτρέψει μια συζήτηση πάνω σε συγκεκριμένους παναμέτρους. γιατί δεν τον σκέφτεστε αυτό. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε στο Κοινοβούλιο. Όπως γνωρίζετε, σε μερικές χώρες μέλη, σε περιφέρειες, οι κυβερνήσεις, οι τοπικές συναρμόδιες με την υγεία, ε, την εκπαίδευση κτλ. Οι κεντρικές κυβερνήσεις ασχολούνται με τις αμυντικές δεπάνες και άλλες παραγωγικές επενδύσεις. Τώρα πρέπει να έχουμε νέα μέτρα εξυγίανση σε διάφορε χώρε. Πιστεύετε ότι η υγεία, η ευημερία, η εκπαίδευση, οι δαπάνε αυτές πρέπει να προστατεύονται όσο γίνεται περισσότερο. Και πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξουν ε, μειώσει αμυντικέ, όπω το Κοινοβούλιο έχει έτσι κι αλλιώ συμπεριλάβει σε έκθεσή του. Και δεύτερον, στην Ισπανία μάθαμε σήμερα ότι υπάρχουν 6,2 εκατομμύρια άνεργοι, νέο ρεκόρ. Ευχαριστώ. Έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, για τα σχόλια και τις ερωτήσεις της κυρίας Ποδηματά. Κατέδειξαν το γεγονός ότι για να υπάρξει απόφαση να παραταθεί ένα πρόγραμμα ή να παραταθεί η περίοδος ε, δημοσιονομικής εξυγένσης χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση από τις χώρες της Ευρωζώνης που παρέχουν εγγυήσεις για τα δάνεια που δίδονται σε αυτές τις χώρες. Και αυτό προϋποθέτει αποφάσεις κάθε κοινοβουλίου χώρας της Ευρωζώνης. Αυτό είναι πολύ συχνά δυσχέρεια για την ε, κατάρτιση πολιτικής. Ξέρετε τα προγράμματα αυτά έχουν σχεδιαστεί ούτω ώστε να λαμβάνουν υπόψη και ανησυχίες για θέματα πολιτικής, δηλαδή τι χρειάζεται για την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική, για την πολιτική απασχόληση, από τη μία, από την άλλη, έχουμε και τους ε, χρηματοδοτικούς περιορισμούς. Και σε κάποια φάση στα πλαίσια των συζητήσεων του Eurogroup πρέπει να ακουστεί και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λαμβάνεται μια απόφαση και πρέπει να ληφθεί ομόφωνα. Και φυσικά τα κράτη-μέλη λαμβάνουν υπόψη και τους χρηματοδοτικούς περιορισμούς. Όσον αφορά την επισκόπηση για την Ελλάδα ή τη συμπερίληψη της Ελλάδας ή κάποιας άλλης χώρας ε, προγράμματος στη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών έχουμε ένα συνεχές πρόγραμμα επιτήρησης στις χώρες προγράμματος που είναι πιο συγκεκριμένο, πιο ακριβές από τη διαδικασία επιτήρησης μέσω της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών. Και επιπλέον έχουμε και αυτές τις τριμηνιαίες επισκοπήσεις. Οι χώρες προγράμματος επιθεωρούνται κάθε τρεις μήνες και αν χρειαστεί τροποποιείται το πρόγραμμα όπως ακριβώς ε, επιμικίναμε το πρόγραμμα ε, δημοσιονομικής προσαρμογής και στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία. Δηλαδή, λοιπόν, εάν τις εντάξουμε και στη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών θα είχαμε επικάλυψη. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι ουσιώδες να διατηρήσουμε την τωρινή πρακτική τριμηνιαίων επισκοπήσεων των χωρών προγράμματος. Ο κύριος Τρεμόζα αναφέρθηκε στις στρατιωτικές δαπάνες. Όπως ξέρετε, στα πλαίσια της κατανομής αρμοδιοτήτων στην Ένωση, οι αμυντικές δαπάνες είναι εθνικό θέμα. Βεβαίω ε, πρέπει να συμμετάσχουν οι δαπάνες αυτές στην δημοσιονομική εξυγίανση. Δεν μπορούν να υπάρχουν οι αγελάδε στην επισκόπηση των δαπανών όταν τα κράτη-μέλη έχουν τόσο ε, σημαντικούς δημοσιονομικούς περιορισμούς. Έχω πλήρη συνέστηση το απαράδεκτο επίπεδο ε, ανεργίας στην Ισπανία. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία η Ισπανία να επανέλθει στην οδό της ανάκαμψης, της βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, θέσεων απασχόλησης. πρέπει να αναθεωρηθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δεν έχει αποκατασταθεί πλήρω, δεν έχει ανακεφαλαιοποιηθεί. Πρέπει να αναλυφθούν και άλλε δράσει, ενεργή πολιτική στην αγορά εργασία, για παράδειγμα, και συνοδευτικά μέτρα για την απασχόληση που να συνδυάζονται για παράδειγμα με το ε, σχέδιο εγγύσεων για την ενεργεία των ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και προσβλέπω και στην επόμενη συνάντηση μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι τελειώνουν και οι εργασίες μας. Θα ξανασυναντηθούμε στις 7 Μαΐου στις 9 το πρωί και μετά από 1.30 μέχρι τις 3 το απόγευμα σε αυτή την αίθουσα για να συζητήσουμε το θέμα της Κύπρου. Στις 8 Μαΐου, όπως είπατε, θα έχουμε εδώ μαζί μας τον Επίτροπο Ρεν, καθώς και εκπρόσωπο της ΕΚΤ για να συζητήσουμε το θέμα της Κύπρου. Δυστυχώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα είναι παρόν, αλλά αργότερα κάποια άλλη στιγμή το Μάιο. Και βεβαίως ε, και κλεισμένων των θυρών. Προσπαθούμε ε, να μην γίνει αυτό στο μέλλον, να αποφευχθεί αυτό, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα επί του παρόντος. Έτσι ώστε να συζητήσουμε θέματα που άπτονται της Τρόικας. Τώρα θα γίνει μια ιδιωτική συζήτηση για τους διαπραγματευτές του SSM, του ενίου εποπτικού μηχανισμού. Θα παραμείνει η διερμηνία για την συνάντηση του SSM.